Παναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά ε, τη χθεσινή ημέρα. Καθώ επίση και τα κείμενα έχουν δημοσιευθεί, υπάρχουν αντιρρήσει όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά. Έχω δύο ανακοινώσει ακόμα